Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Welcome to this meeting Καλώς ορίσατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Πρώτο σημείο η έγκριση της ημερήσιας διάταξης να σας πω ότι θα αναβληθεί το σημείο 8 και το σημείο 13 θα συζητηθεί αμέσως μετά το σημείο 14. Υπάρχουν ε, ε, στάσεις, προτάσεις, δεν βλέπω κάποιον, επομένως εγκρίνεται η μερίσια διάταξη και πάμε στο σημείο 2, ανταλλαγή απόψεων για την τριδιάστατη εκτύπωση, μια νέα πρόκληση στον τομέα των ε, ε δικαιωμάτων ε, ιδιωτικής ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και τις αστικές ευθύνες και να δώσω το λόγο αμέσως στην κυρία Μπερζερόν, την εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να σας υπενθυμίσω λίγο την τρισδιάστατη τεχνολογία για να μπορέσουμε να είμαστε και σαφείς ως προς τα όσα θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Η τρισδιάστατη εκτύπωση εμφανίστηκε στο τέλος της δεκαετίας του 80 αλλά χάρη στην ε, μεγάλη πρόοδο και ταχεία πρόεδρος της τηλετεχνολογίας ε, έγινε πιο προσβάσιμη και πιο προσιτή ε, για χρήση σε καθημερινό επίπεδο χρησιμοποιείται από τον κλάδο εδώ και 30 χρόνια χωρίς να δημιουργήσουν νομικά προσκόμματα για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχουν ρυθμιστεί αυτά, ρυθμίζονται συνήθως μέσω συμβάσεων. Και επίσης το δίκτυο των επαγγελματιών που παράγουν βιομηχανικά ή σχεδόν βιομηχανικά προϊόντα τα οποία ε, θα μπορούσαν να παράγουν μία σειρά ε, ε, προϊόντων για να τα πουλήσουν ε, επειδή ακριβώς είναι δαπανηρή η διαδικασία των τρισδιάστατων εκτυπώσεων δεν, προσφέρει, δεν δημιουργεί προβλήματα. Το πρόβλημα είναι όταν αρχίζουν να το χρησιμοποιούν καθημερινοί άνθρωποι. Η εκθετική αύξηση της τεχνολογίας αυτής στον κόσμο της τεχνολογίας μας οδήγησε σε ένα φαινόμενο εκμοκρατισμού της χρήσης των τριδιάστατων εκτυπώσεων. Έτσι μπορούμε να έχουμε ένα πανομοιότυπο αντίγραφο από πολλαπλές πηγές οι οποίες είναι εύκολα προσβάσιμες ή μέσω διαδικτύου ή μέσω ε, τρισδιάστατων ε, σαρωτών. Ε, τίθεται λοιπόν θέμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα ε, δημιουργού, δικαιώματα ευρωσιτεχνίας κλπ. Ε, ακόμα και η μερική αναπαραγωγή ενός έργου χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού υπάρχει περίπτωση ε, να διαδοθεί επίσης και μέσω διαδικτύου, για παράδειγμα λογισμικού. Αυτά όλα είναι παραποίηση. Ε, όλες οι ε, εκτυπώσεις σε τρισδιάστατο επίπεδο όμως δεν είναι συστηματικά παράνομες και όλες οι διαδικασίες δεν είναι απαραίτητα ε, παραποίηση. Η τρισδιάστατη εκτύπωση που γίνεται σε ιδιωτικό επίπεδο από απλούς πολίτες και όταν ο σκοπός δεν είναι η εμπορική χρήση, δεν είναι ε, Είναι σαν να εκτυπώνει κάποιο μία σελίδα στον εκτυπωτή του. Αυτά λοιπόν που κάνουν οι ιδιώτε στο σπίτι τους ε, ε, ακόμα δεν είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένα αυτή τη στιγμή διότι οι δυνατότητες των συσκευών που πολλούνται σε προσιτέ τιμέ ε, και αυτό σημαίνει κάτω των χιλίων ευρώ είναι πολύ περιορισμένες. Ε, αλλά η τεχνολογία προχωρά αρκετά γρήγορα. Αυτή τη στιγμή έχουμε απλώς ε, τρισδιάστατα μικροαντικείμενα, κάποιες φιγούρες. Ε, δεν χρησιμοποιείται και ρητίνη από τους ιδιώτες νομίζω και επομένω η χρήση είναι περιορισμένη. Έχουμε λοιπόν και κάποιες πλατφόρμες που λέγονται Fab Labs που χρησιμοποιούνται από ιδιώτες που κάνουν τρισδιάστατες εκτυπώσεις ε, και υπάρχουν και αρκετές πλατφόρμε όμως που χρησιμοποιούν επαγγελματίε. Πέραν όσον αφορά το γεγονό ότι υπάρχει ε, και ε, απώλεια εισοδημάτων, υπάρχουν και δεντολογικά ζητήματα, κυρίως στο δικαίωμα στην ακαιρεότητα του έργου του δημιουργού, μπορεί να παραβιαστεί επειδή προσφέρεται στο διαδίκτυο πολύ ελεύθερα η δυνατότητα να παράγονται τέτοια ψηφιακά. Ε, μας ενδιαφέρουν επίσης ε, ε κυρίως τα θέματα πνευματικής διοκτησίας. Δεν θα πρέπει όμως να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένους κλάδους ε, και ούτε και στους ιδιώτες. Με ενδιαφέρει κυρίως, για παράδειγμα, ο τομέας ε, της ιατρικής και το διοντολογικό πρόβλημα που προκύπτει. Διότι διάβασα ότι μπορούμε σχεδόν να ε, εκτυπώσουμε ανθρώπινο δέρμα. Το πρόβλημα είναι αρκετά περίπλοκο, διότι υπάρχει το θέμα της πνευματικής διοκτησίας ε, των τρισδιάστατων εκτυπώσεων και τα θέματα της αστικής ευθύνη ε, για ένα ελαττωματικό προϊόν, το οποίο θα μπορούσε να συμβεί πολύ συχνά στο μέλλον. Τα θέματα επίσης ε, των πνευματικών δικαιωμάτων της λογοτεχνικής δημιουργίας επιτρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των παράνομων τρισδιάστατων εκτυπώσεων. Τώρα, εάν είναι ελαττωματικά τα προϊόντα, εκεί υπάρχουν προβλήματα σε θέματα νομικής. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε το δημιουργό ε, του ε, φακέλου CIA που είναι οι μακέτες πληροφορικής. Αλλά επίσης μπορεί να υπάρχει τρισδιάστατη εκτύπωση κατά παραγγελία. Ε, να υπάρχει ο αγοραστής ο οποίος θα μπορούσε να είναι υπεύθυνο. Ε, η πλατφόρμα διάδοσης πληροφοριών για τα ε, θέματα αυτά της διαδικτυακής εκτύπωσης και πολλοί άλλοι. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα ε, προϊόντα τα οποία παράγονται με τρισδιάστατη εκτύπωση ε, πληρούν προϋποθέσεις ασφαλείας και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται από ιδιώτες δεν είναι τοξικά, είναι ανθεκτικά στη θερμότητα κλπ. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα τα οποία παράγονται τρισδιάστατα από ιδιώτες ε, είναι σωστά. Ποιος είναι υπεύθυνο σε περίπτωση ατυχήματο και ποιο είναι υπεύθυνο για τα ελαττωματικά προϊόντα. Ο παραγασκευαστής, ποιος είναι ο κατασκευαστής σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής ο οποίος εκτυπώνει μόνος του ένα προϊόν από μία σελίδα την οποία έχει εκτυπώσει από το διαδίκτυο, είναι ο κατασκευαστής ή είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε το πρόγραμμα. Όλα αυτά δημιουργούν λοιπόν κάποια προβλήματα τα οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να μας βοηθήσουν να βρούμε κατάλληλη ρύθμιση για τα τρισδιάστατα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να ανακόψουμε την πορεία των καινοτομιών, ίσα ίσα να τις βοηθήσουμε και να προλάβουμε τυχόν προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να μην υπάρξει παραποίηση συστηματικά και η δική μας η αποστολή είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους αλλά και όλους τους πελάτες ε, πιθανών ε, των τρισδιάστατων προϊόντων για να αντιμετωπίσουμε πιθανούς κινδύνους για την παρασκευή και χρήση προϊόντων τα οποία εκτυπώνονται μέσω αυτού του συστήματος. Ελπίζω να με βοηθήσετε διότι εγώ δεν έχω καταφέρει να δω όλους τους τομείς αυτού του ε, θέματος και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Mr. De Grandes. Ο κύριος Δεκράντες Πασκουάλ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για αυτή την πρώτη ενημέρωση ε, για το θέμα αυτό, ε, για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, ε, ιδίω σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Είναι αναπόφευκτο να μην αρχίσουμε να συζητάμε για ρομπότ, για τρισδιάστατα και για τις ε, παρισφρήσεις της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας. Ε, σήμερα σε όλα ε, τις εφημερίδες του κόσμου αναφέρεται το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς λοιπόν ως Ευρωβουλευτές έτσι το βλέπουμε και πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα στην έκθεση αυτή να ε, αναπτύξουμε το θέμα, διότι πρόκειται για μια νέα τεχνολογία. αυτέ οι τρισδιάστατε εκτυπώσεις είναι νέα τεχνολογία και πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ρύθμιση. Υπάρχουν αρκετοί κλάδοι που τις ε, χρησιμοποιούν σοβαρά και υπάρχουν σοβαρές δυνατότητες ε, μεγάλων κερδών. Ε, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελεί πραγματική επανάσταση στην καθημερινή ζωή και κατά την άποψή τους ε, θα είναι μια αγορά η οποία έχει δυνατότητες πολύ μεγάλης ανάπτυξης στα μελλοντικά χρόνια. Ε, πρέπει να δούμε όμως τι θα γίνεται στην έκθεση. Η αποστολή μας είναι να συζητήσουμε και να λύσουμε τις συνέπειες που υπάρχουν για τους κείμενους κανόνες σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις βασικές προκλήσεις. Δικαιώματα δημιουργού, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ε, και ε, επαγγελματικά σήματα. Επίσης, εμπορικά σήματα. Θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται. Μπορεί να υπάρξει και μια μαύρη αγορά κλωνοποιημένων και ε, τρισδιάστατων προϊόντων και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα με βάση κάποια κριτήρια. Καταρχάς, πρώτον θα πρέπει να αποφύγουμε οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις να παραβιάσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάποια νομικά θέματα που τίθενται είναι η ε, μεταφόρτωση τρισδιάστατων προϊόντων ε, παρά την ε, θέληση του δημιουργού και τι θα γίνει με τα παραποιημένα προϊόντα τρισδιάστατα. Επίσης, οι εκτυπωτές αυτές μπορούν να παράξουν οποιοδήποτε προϊόν, όπως για παράδειγμα και παράνομα προϊόντα, ναρκωτικά ή όπλα. Ε, λέγεται ότι κυρίως χρησιμοποιούνται για την ιατρική, για προσθετικά μέλη, αλλά αυτά τα προϊόντα υπόκεινται σε πολύ αυστηρή ε, νομοθεσία βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Εάν κάποιος λοιπόν μπορεί να εκτυπώσει ένα προϊόν ε, στο σπίτι του και υπάρχουν ελαττωματικά προϊόντα λόγω προβλημάτων στην εκτύπωση, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη. Δεύτερον, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο για τι τρισδιάστατες εκτυπώσεις που να λύνουν και τα θέματα της ευθύνη από νομική ε, τα προβλήματα για την ευθύνη ε, για τα προϊόντα αφορά τον κατασκευαστή ω υπεύθυνο για τα ελαττωματικά προϊόντα κατά τη χρήση των προϊόντων. Αλλά όταν ο πελάτη είναι και ο κατασκευαστή του προϊόντος στο σπίτι του μπορεί να υπάρχουν και κάποιες ε, παρενέργειες. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι όσα υπάρχουν, θα υπάρξουν σε θέματα τρισδιάστατων εκτυπώσεων θα πρέπει να σέβονται και την κείμενη νομοθεσία σε θεμελιώδη δικαιώματα και πνευματικά δικαιώματα. Πρόκειται για ένα καινοτόμα τομέα και από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε. Σήμερα απλώ ε, θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, αλλά μα περιμένει στη συνέχεια ε, μια εντυπωσιακή δουλειά και πιστεύω ότι μπορούμε με τη συνεισφορά όλων να καταφέρουμε αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας να θέσει τα θεμέλια μελλοντικής νομοθεσίας ε, όπως πρέπει και όπως μας υποχρεώνει ούτως ή άλλως και το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα και πραγματικά αντιμονώ να συνεργαστούμε. Εγώ βασικά έχω μεγάλη σχέση με την τεχνολογία και βλέπω πάντοτε τα τεράστια πλεονεκτήματα που μας φέρνει, που δεν είναι τόσο καινούργια μεν, αλλά είναι ευθυνά πια ε, αυτή τη ριζιάστατη τεχνολογία εκτύπωσης η οποία ε, θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί μέσα από αυτό το νέο νομικό πλαίσιο. Μπορούν να γίνουν πολλά στον περιβαλλοντικό τομέα για παράδειγμα για να μειώσουμε το κόστος μεταφοράς, για γρήγορη ανάπτυξη Νέων προϊόντων, ας πούμε βελτιωμένα ηλιακά πάνελ ε, και τα λοιπά. Φυσικά, έχουμε και πολλά νομικά ζητήματα και προκλήσεις ε, δύσκολες μπροστά μας. Ας πούμε, ο, νόμος ε, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή για τα πνευματικά δικαιώματα που δεν ε, συμβαδίζουν με, τα, με τους φθηνούς αυτούς εκτυπωτές για τρισδιάστατη εκτύπωση, οπότε πρέπει να βρούμε λύση για αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, θα μπορεί ο κόσμος να κατασκευάσει πιστόλια στο σπίτι του. Αυτό είναι μία από τις προκλήσεις ε, που ενέχει η τεχνολογία. Φυσικά υπάρχει και το θέμα της ευθύνης. Πραγματικά με ενθουσιάζει αυτό το θέμα και περιμένω με αδημονία πότε θα ε, προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλα υπόθηκαν για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ήθελα να πω σε όλους ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό, πολλές δυνατότητες με αυτή τη νέα τεχνολογία και επειδή μας ε, ενδιαφέρει η καινοτομία και η πρόοδος, ε, δεν θα φρενάρουμε αυτή την εξέλιξη. Όμως πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας και τους κινδύνους που ενέχει. Εμείς βέβαια περιεραζόμαστε σε νομικά ζητήματα, το θέμα της διανοητικής ιδιοκτησίας και μπορούμε να εμπνευστούμε από τις υφιστάμενες αρχές. Όμως γενικά υπάρχει το θέμα της ευθύνης. Ε, αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι θα έχουμε σύντομα στην αγορά τρισδιάστατες εκτυπώσεις πάρα πολύ φθηνές, οι οποίες ε, ε, πραγματικά θα φέρουν στην αγορά φθηνά προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να δούμε ζητήματα εγκρίσεων, τυποποίησης, ε, γιατί μπορεί τελικά με τους εκτυπωτές ε, αυτούς να έχουμε αλλατοματικά προϊόντα που βλάπτουν την υγεία. Είναι κίνδυνος αυτό. Άρα, πώς θα προχωρήσουμε στο θέμα των εγκρίσεων, της ε, εμπορικής χρήσης αυτών των προϊόντων πώς θα φτιάξουμε αλληλέγγυες οικονομίες, γιατί μιλήσαμε για τη βιομηχανία και για το άτομο. Και υπάρχει η συνεργασία μεταξύ των δύο. Κάποιος φτιάχνει ένα προϊόν, το δίνει στο φίλο του, αυτό συνεχίζει να το εξελίσσει. Δεν ξέρουμε τελικά ε, ποιος είναι ο αρχικός εμπνευστής. Είναι το η λεγόμενη shared economy είναι σημαντικό να τα έχουμε αυτά στο μυαλό μας όταν μιλάμε για αυτή τη τεχνολογία και νομίζω ότι είναι όμως ένα εξαιρετικό θέμα. Σου εύχομαι, Ζωέλ, να έχεις μεγάλη έμπνευση. Ο κύριος Φως. Ευχαριστώ. Κατά βάση, όπως είπαν και οι υπόλοιποι, στην ίδια κατεύθυνση να πω και εγώ ότι έχουμε τώρα ε, κάτι καινούριο, ε, αλλά δεν εκτυπώνουμε σπίτια, ε, εκτυπώνουμε συσκευές ή ξέρω εγώ νεφρά. Είναι πράγματα που μας δίνουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουμε με διάφορες μορφές, αλλά μπορούν να φέρουν μια επανάσταση στη ζωή μας γενικότερα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της ευθύνης εδώ. Υπάρχει μια βάση, ήδη έχουμε μια έκθεση για τη ρομποτική και ήδη ε, έχουμε κάποια γνώση, όμως πρέπει να διαφοροποιηθούμε. Πρέπει να δούμε, για παράδειγμα, ποιος θα είναι υπεύθυνος τελικά για αυτό το προϊόν. Υπάρχουν ε, ψηφιακά δεδομένα που ε, υφίστανται ήδη και γι' αυτά υπάρχει κάποια ευθύνη. Αν είναι, ας πούμε, ελαττωματική μια συσκευή που επεξεργάζεται ψηφιακά δεδομένα ή αν η χρήση της είναι ελαττωματική. Πώς γίνεται. Θα πρέπει τέλος πάντων να βασιστούμε σε αυτά, αλλά κάνουμε και μια διαφοροποίηση σε επίπεδο διανοητικής ιδιοκτησίας, πατέντας Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο, αλλά στην πράξη είναι λίγο δύσκολο. Τι γίνεται όταν κανείς ε, ε, εκτυπώνει στο σπίτι, αν έχει πολύ ζέστη θα λιώσει, ας πούμε, το προϊόν. Τι γίνεται με τα υλικά, πώς τα προμηθεύεσαι. Η ευθύνη είναι πολύ σημαντική, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να κοιτάξουμε. Το σημαντικό είναι να διαφοροποιήσουμε με βάση τον τομέα στον οποίο ενδιαφερόμαστε. Would the Commission wish to take the floor? Μήπως θέλει η Επιτροπή να λάβει το λόγο. Ναι, σας ευχαριστούμε. Κάτι βιέκτου από τη Γενική Διευθύνση ε, τα θέματα καταναλωτή. Καλωσορίζουμε ορίζουμε στη συζήτηση που γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντική και επίκαιρη γιατί διαπιστώνουμε ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και από την βιομηχανία αλλά και από ιδιώτες. Αναφέρθηκε και ως ορθά η σημασία των πλατφορμών που έχουν δημιουργηθεί για τη συνεργασία και αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν ζητήματα για τον τομέα της αστικής ευθύνης, για τον τομέα των συμβάσεων. Γιατί δημιουργούνται ερωτήματα. Για παράδειγμα, δεν είναι ξεκάθαρο ποιο είναι ο πολιτή σε μια τέτοια εικονική ε, πλατφόρμα συνεργασία. Και επίση δεν μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο τι ακριβώ έχει αγοράσει ο πελάτη. Ε, στην περίπτωση όπου πωλείται μια μακέτα τρισδιάστατης εκτύπωσης, αυτό που έχει αγοραστεί είναι το προϊόν ή μόνο το αρχείο, ε, το σχεδιαστικό τον Δεκέμβριο του 2015 η Επιτροπή έχει ε, υπέβαλε μια ε, πρόταση οδηγίας για τους παρόχους ψηφιακού περιεχομένου που καλύπτει και τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες έχει παρασχεθεί ε, προβληματικό ψηφιακό περιεχόμενο και καλύπτεται η αποζημίωση των καταναλωτών. Ένα αρχείο υπολογιστή για ψηφιακή εκτύπωση αποτελεί παράδειγμα ψηφιακού περιεχομένου που θα καλυπτόταν, που, καλύπτεται από αυτή την οδηγία. Αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλα ζητήματα πολύ σημαντικά, συναφή, που έχουν σχέση με το δίκαιο αδικοπραξίας, όπως η πρόκληση ζημίας, η ή άλλα που περιπλέκονται ακριβώ επειδή η αλλα που περιπλεκονται ακριβως επειδη η αλυσιδα των παραγωγών και των πελατών σε αυτού του τύπου τις ε, συναλλαγές είναι πολύ ε, μακρά. Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε ή να συζητήσουμε αυτά τα περίπλοκα ζητήματα. Είναι παρόν και ένας ε, συνάδελφος ο οποίος θα μπορούσε να σας δώσει λίγες περισσότερες πληροφορίες για το ζήτημα της αστικής ευθύνης. Γενική Εσωτερικής Αγοράς. Καλωσορίζουμε και εμείς την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πράγματι, η διάστατη εκτύπωση δημιουργεί ε, ερωτηματικά. Είναι μια πρόκληση, όπως είπε και η συνάδελφος Κάτια. Γιατί δημιουργεί, μεταβάλλει μάλλον, αλλάζει την παραδοσιακή ε, λειτουργία του παραγωγού και τη σχέση του με τον διανομέα και τον τελικό καταναλωτή. Αλλάζει αυτή η αλυσίδα και δημιουργούνται νέες προκλήσει τι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ένα σημαντικό ε, νομοθετικό εργαλείο είναι η οδηγία για την αστική ευθύνη για τα προϊόντα από το 1985 την οποία έχουμε ξεκινήσει να αναθεωρούμε. Έχει ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση για να δούμε αν συνεχίζει να εκπληρώνει τον σκοπό της. Και προσβλέπουμε να ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση μέχρι τέλο τη χρονιά. Η ψηφιακή εκτύπωση και αυτέ οι εξελίξει τεχνολογικέ είναι μέρο τη αξιολόγηση, τι λαμβάνουμε υπόψη μα. Γι' αυτό λοιπόν ε, ε, προσβλέπουμε στη συνεργασία με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί τη έκθεση αυτή για να διαπιστώσουμε ε, όλα τα προβλήματα, όλε τι προκλήσει που έχουν δημιουργηθεί από την τρισδιάστατη εκτύπωση και ιδιαίτερα όσον αφορά την αστική ευθύνη για τα προϊόντα. Θα ήθελα επίση να δώσω στο λόγο ε, στον συνάδελφο για να μας ε, μιλήσει λίγο για το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ακούτε τους εκπροσώπους της Επιτροπής τον ένα μετά τον άλλον. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για το, την πνευματική ιδιοκτησία, όπως ε, η συγγήτρια σωστά ανέφερε. Το υφιστάμενο σύστημα για την προστασία τη πνευματική ιδιοκτησία είναι πράγματι πολύ ε, λειτουργικό και ορθό. Βεβαίω χρειάζεται κάποιε μικρέ ε, τροποποιήσεις για να ανταποκριθούμε στι αλλαγέ που έχει φέρει αυτή η τεχνολογία. Αυτή η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ γρήγορα και δεν γνωρίζουμε ακόμα πού θα καταλήξουν τα πράγματα. όπω πολλοί συνάδελφοι ε, πολλοί, πολλοί, πολλά μέλη του, του Κοινοβουλίου είπαν ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε την καινοτομία και όχι να την μπλοκάρουμε. Επομένω, οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να γίνει προ αυτή την κατεύθυνση. Εμεί από την πλευρά μα ε, παρακολουθούμε τι εξέλιξει στην αγορά για να δούμε πώ επηρεάζεται το δίκαιο πνευματική ιδιοκτησία, τι συμβαίνει με τα παραποιημένα προϊόντα, τα... και όπως σωστά είπε και η συγγήτρια, αλλάζει το business model, αν θέλετε, το, το τρόπος λειτουργίας εκείνων που δημιουργούν προϊόντα μαϊμού. Εξαιτίας και χάρη αυτής της χρήσης της, της εκτύπωση. εκτύπωσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Μήπως η συγγήτρια θέλει το λόγο για να κλείσει. Η συγγήτρια δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Πράγματι το ζήτημα είναι μεγάλο και είναι ευχάριστο το ότι ζούμε σε μια εποχή τεχνολογικών εξελίξεων και γενοτομιών έχουμε τη δυνατότητα εδώ να νομοθετήσουμε όλοι μαζί και με τη βοήθειά σα και με, τα φώτα της που θα μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη τις γνώσεις της, ε, να νομοθετήσουμε λοιπόν ήδη από την αρχή ε, αυτά τα ζητήματα που δημιουργούνται με τη τρισδιάστατη εκτύπωση ε, και να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα στην ρίζα του, από την αρχή πριν υπάρξουν οποιαδήποτε ε, προβλήματα ή ατυχήματα. Μπορούμε να κλείσουμε, λέει ο Πρόεδρος, αυτό το σημείο τη σημερινή διάταξη. Θα περάσουμε στο σημείο 3, την ακρόαση και θα δώσω ε, στον κύριο Καβαντά το λόγο για να προεδρεύσει στην ακρόαση.